Ψηφίσουμε τα 7 ψηφίσματα. Τώρα έληξε η συζήτηση. Θα εξετάσουμε τα ψηφίσματα τώρα. Επόμενο θέμα. Ψηφίζουμε τα 7 ψηφίσματα για την Ζιμπάμπουε. Το κοινό ψήφισμα 7 πολιτικών ομάδων. Παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, τροπολογία αριθμός 1. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές να το ελέγξουμε καλύτερα. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά λοιπόν την τροπολογία αριθμός 1. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αιτιολογική αναφορά 6. Η κυρία Γκόμες θέλει μια προφορική τροποποίηση να προτείνει. Παρακαλώ κυρία Γκόμες, μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Προτείνω εκεί που αναφερόμαστε στην Αφρικανική Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων Τολών που έχει στην υπογράψη και η Ζιμπάμπουε, λέει το κείμενο τώρα, which Zimbabwe is a full member, είναι μέλος, να βάλουμε που έχει επικυρώσει Zimbabwe καλύτερα. Δεν βλέπω να έχει κανείς αντίρρηση για την προφορική αυτή τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε το κοινό ψήφισμα στο σύνολό του. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, ψήφισμα για την Βενεζουέλα. Κοινό ψήφισμα. Το ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. And now the... Και τώρα Ψήφισμα για τη Βόρεια Κορέα. Καταρχήν παράγραφος 2. Κατά τμήματα ψηφοφορία, παρακαλώ. Για το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Κατά τμήματα ψηφοφορία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα το σύνολο του τροποποιημένου ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία όμως. Παρακαλώ, ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίστε. The vote is της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. I have a of Έχω κάποιες ανακοινώσεις να κάνω. Από την ομάδα του ΕΛΚΑ μου έχει ζητηθεί να ορίσουμε την Ελίζα Μωρίν Τσάρτιερ ω μέλο τη Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Δύο Φύλων. Σχόλια από αυτού. Ο ορισμό λοιπόν εγκρίνεται. Επίση από τι